Αγαπητοί συνάδελφοι, <laughs> με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να καλωσορίσω δύο υπουργού από τη Μαλτέζικη Προεδρία, τον κύριο Μπονίτσι που είναι Υπουργό Δικαιοσύνη, Πολιτισμού και Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον κύριο Κρίσιαν Καρντόνα που είναι Υπουργό Οικονομικών, Επενδύσεων και Μικρών Επιχειρήσεων. Καλώ ήρθατε κύριε Υπουργή στην Επιτροπή μα. Κύριε Μπονίτσι, θα λάβετε εσείς πρώτος το λόγο, θα μας κάνετε την παρουσίασή σας και θα ακολουθήσουν ερωταπαντήσεις. Κύριε Υπουργέ Μπονίτσι, έχετε το λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά κυρία Πρόεδρε. Η Ευρώπη θεωρώ, θεωρείται υπόδειγμα ευημερία, ανάπτυξης και ειρήνης. Και αυτό το σημαντικό επίτευγμα υλοποιήθηκε χάρη στο ευρωπαϊκό όραμα και παρά τις, τους ενδιασμούς πολλών για το κατά πόσο η συνθήκη του Μάστρικ θα τελεσφορήσει και θα συνεργαστούμε στενά και κατά την 60η επέτειο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου ε, Ήρθε η σειρά της Μάλτας για να ασκήσει την Προεδρία. Νιώθουμε μεγάλο προνόμιο λοιπόν, τιμή και ευκαιρία, τη δυνατότητα να προεδρεύσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα πρέπει να, από... να εξετάσουμε από κοινού την παρακαταθήκη των τελευταίων 60 ετών και να ε, ενημερώσουμε τους πολίτες μας για τα ωφέλη αυτού του σχεδίου, γιατί μερικές φορές ξεχνούν τα πλανεκτήματα του Ευρωπαϊκού Σχεδίου. Θα έχουμε λοιπόν μια καλή ευκαιρία για να δώσουμε μια νέα όθηση στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο. Οι πρόσφατες εξελίξεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξαν κατάφορα την ανάγκη να φέρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της, με μια καλύτερη επικοινωνία για τα μέτρα που λαμβάνονται και να εξηγήσουμε καλύτερα στους συμπολίτες μας ότι με το έργο μας εξυπηρετούμε τους πολίτες και τους επιτρέπουμε να υλοποιήσουν τις επιθυμίες τους και τις φιλοδοξίες τους. Οι πολιτικές εξελίξεις του τελευταίου χρόνου μας στιγμάτισαν και η ανάγκη για μεταρρύθμιση είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Και μάλιστα ε, σήμερα είναι ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη του να έρθουμε πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες. Τα γεγονότα της τελευταίας χρονιάς έχουν ε, συγκλονίσει στη θέμελα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και η Μάλτα θέλει να συμβάλλει με το λιθαράκι της στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο και στην ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς στο Συμβούλιο αλλά και εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μεριμνήσουμε ώστε να δοθεί αυτή η όθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχυθεί. Φυσικά ένα εξάμεινο είναι ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά είμαστε φιλόδοξοι και θέλουμε να συμβάλλουμε στην πρόθεση του προγράμματός μας για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο αξιόπιστη. Κανένας βέβαια δεν έχει ψευδεστήσεις ε, ούτε παραλυρήματα μεγαλείου. Γνωρίζουμε τους περιορισμούς, αλλά ε, έχουμε ξεκάθαρη την πορεία μας και ξέρουμε τι θέλουμε. Θέλουμε να συνεργαστούμε στενά, με ειλικρίνεια και με διαφάνεια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ε, ήταν πρώην Ευρωβουλευτές. Οπότε θα καταλάβουμε καλύτερα την σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν εξοικειωμένοι με το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εσείς είστε οι άμεση εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών και θα μας βοηθήσετε ώστε να νομοθετούμε υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή θα είναι ο βασικός μας μύτος της Αριάδνης. Έτσι θα καταφέρουμε να δώσουμε μια νέα όθηση στο έργο μας και να φέρουμε τους συμπολίτες μας πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και καταλήξαμε σε έξι προτεραιότητες. Στη μετανάστευση, την ασφάλεια, την εσωτερική αγορά, την πολιτική γειτονία, την κοινωνική ένταξη και τα ναυτιλιακά θέματα. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας. Γιατί οι συμπολίτε μα ε, έχουν πολύ σοβαρέ ανησυχίες και εύλογε και θα πρέπει να του αφογκραστούμε. Ο Πρωθυπουργό μα, όταν έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την επόμενη εβδομάδα συγκεκριμένα στην Ολομέλεια, θα έχει την ευκαιρία να σα αναπτύξει πιο λεπτομεριακά το πρόγραμμα τη Μαλτέζικη Προεδρία. Οπότε, με την άδειά σα, ε, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σα ε, πω λίγα λόγια για το πρόγραμμα εργασιών ε, της Μαλτέζικης Προεδρίας και μάλιστα στα αγγλικά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που δώσατε το παρόν σήμερα το απόγευμα. Είναι τιμή και για μένα και για τον φίλο Υπουργό Καρντόνα που βρισκόμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το θεσμικό όργανο που συνδέεται ε, άρρηκτα με τους πολίτες. Και Γι' αυτό νιώθουμε ιδιαίτερα υπόλογοι προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο τομέας της δικαιοσύνης είναι ένας τομέας που μείνει είναι ιδιαίτερα προσφυλής, αλλά και στους συναδέλφους το ίδιο, γιατί περισσότεροι είμαστε δικηγόροι στο επάγγελμα και πιστεύουμε ότι ο τομέας της δικαιοσύνης συνδέεται άρρηκτα με τις ε, πιο θεμελιώδεις ε, και βασικές ε, ελευθερίες και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σεβασμό της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου. Και όπως προβλέπει και η ίδια συνθήκη, αυτές είναι οι αξίες ε, που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Πρώτη φορά η Μάλτα θα ασκήσει αυτή την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση και να σημειώσουμε πρόοδο σε όλα τα θέματα των προτεραιοτήτων μας. Γιατί για πολλά χρόνια είμαστε η γέφυρα μεταξύ διαφόρων πολιτισμών. Ακόμα και η γλώσσα μας είναι ένα συνοθήλευμα διαφορετικών πολιτιστικών στοιχείων. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είμαστε ιδιαίτερα επιρρεπείς προς τη συνεργασία και αυτό το εξάμεινο που θα ακολουθήσει θα εξασφαλίσουμε, θα φροντίσουμε τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε την αγαστή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βασική μας προτεραιότητα είναι σαφής. Οι προτεραιότητες μας μάλλον είναι ξεκάθαρες. Δεν υπάρχουν ιστεροβολίες ούτε ε, κρυφές προθέσεις. Θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο στις νομοθετικές προτάσεις που βρίσκονται στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Προτάσεις ε, για τα, τις συμβάσεις, ε, το ηλεκτρονικό περιεχόμενο και τις ηλεκτρονικές αγοροπολισίες. Ενδιαφέροντα θέματα για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, που περιμένουμε ενδιαφέρον την πρόοδο στις συζητήσεις αυτές. Οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο ε, προβλέπουν κυρίως ε, την εξέταση της πρότασης για το ψηφιακό περιεχόμενο. Το Συμβούλιο Δικαιοσύνη και Ιστορικών Υποθέσεων του περασμένου Δεκεμβρίου είχε μια συζήτηση πολιτική γύρω από τρία θέματα το ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο, άλλα δεδομένα και ισορροπία μεταξύ της των, ε, υποκειμενικών και των κριτηρίων υποκειμενικής και αντικειμενικής συμμόρφωσης. Και θα πρέπει να γίνει ακόμη πολύ έργο σε τεχνικό επίπεδο. Πάντως, έχουμε θέσει ήδη το φιλόδοξο στόχο να καταλήξουμε σε μια γενική προσέγγιση για την πρόταση του ψηφιακού περιεχομένου μέχρι το πέρας της Προεδρίας μας. Θα προσπαθήσουμε επίσης να προωθήσουμε το έργο, την πρόταση για τις πωλήσει εμπορευμάτων αγαθών και να εξετάσουμε κατά πόσο το πεδίο εφαρμογή θα πρέπει να παραταθεί, να επεκταθεί και σε πωλήσει offline που γίνονται πρόσωπο με πρόσωπο δηλαδή. το βασικό θέμα των συζητήσεων στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το ίδιο. Γι' αυτό και παρακολουθούμε προσεκτικά τις συζητήσεις στην Επιτροπή Γιούρη και ΙΜΚΟ. Και ελπίζουμε ότι οι εργασίες κατά τη Μαλτέζικη Προεδρία στο θέμα αυτό θα στρώσουν το δρόμο για μια συμφωνία της πρώτης, σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης θα ξεκινήσουμε ε, συζήτηση με την πρόσφατη πρόταση για την αφαιρεγκαιότητα των επιχειρήσεων. Έτσι θα επιτρέψουμε σε βιώσιμες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση να διασωθούν και θα επιτρέψουμε και σε έντιμους επιχειρηματίες να λάβουν μια δεύτερη ευκαιρία. Η πρόταση αυτή περιέχει ένα ε, στοιχείο σημαντικό που αφορά και την κεφαλαγορά και την Ένωση Κεφαλαγόρων και την ε, ενιαία στρατηγική για την ε, ενιαία αγορά. Θέλουμε να μειώσουμε τα εμπόδια των διασυνοριακών επενδύσεων ώστε να ενισχύσουμε την οικονομία μας και να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις προκειμένου να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Η Μαλτέζικη Προεδρία θεωρεί ότι η πρόοδος ε, ε, για τις, στις διαπραγματεύσεις για την αφαιρεγγιότητα, την αναδιάρθρωση και τη δεύτερη ευκαιρία, ε, όλες αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς στο Συμβούλιο. Στόχος μας είναι να γίνει αποτελεσματική συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο στο Συμβούλιο. Και μάλιστα έχουμε δεσμευθεί να αφιερώσουμε νέα εργάσιμες μέρες στο θέμα αυτό. Επίσης, περιμένουμε με μεγάλη αδημονία τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη νέα πρόταση και προσβλέπουμε σε καρποφόρα συνεργασία μαζί σας. Οι συζητήσεις ε, θα συνεχιστούν και επί της ε, προτάσεως αναθεώρησης ε, του κανονισμού των Βρυξελών 2α. Ένας ιδιαίτερα προσφυλή σε ένα κανονισμός, γιατί πιστεύω ότι αυτός ο κανονισμός μπορεί να απλουστεύσει, να διευκολύνει τη ζωή των συμπολιτών μας γιατί επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητά τους. Θα συνεχίσουμε λοιπόν το αξιόλογο έργο της Σλοβακικής Προεδρίας και να προωθήσουμε και το κρίσιμο θέμα των οικογενειακών θεμάτων. Θέλουμε ε, και συζήτηση επί της πολιτικής στο Συμβούλιο Εσωτερικό και Δικαιοσύνης τον Ιούνιο. Γνωρίζουμε ότι τα οικογενειακά θέματα και το ζωτικό συμφέρον του παιδιού είναι θέματα προσφυλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γι' αυτό και περιμένουμε με ανυπομονησία τη σχετική σας γνωμοδότηση. Ε, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό και το θέμα της καταπολέμησης της βίας λόγω φύλου και θα αφιερώσουμε ε, πολλές συζητήσεις στην οριστικοποίηση της πρότασης της Επιτροπής και της απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Και για τα θέματα αυτά θα συνεχίσουμε το έργο των προηγούμενων Προεδριών. Η Μαλτέζικη Προεδρία προτίθεται να οργανώσει και μία διάσκεψη σε εθνικό επίπεδο για την ε, ρητορική μίσους, ένα φλέγον ζήτημα αυτή τη στιγμή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ευελπιστώ ότι θα, με, θα μας στηρίξετε γιατί το πρόγραμμα μας είναι φιλόδοξο και απαιτητικό αλλά είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο χάρη των πολιτών μας, των επιχειρήσεών μας και της κοινωνίας μας ολόκληρης. Και εν κατακλείδη θα ήθελα να διατρανώσω και πάλι την αποφασιστικότητά μας να ενεργήσουμε ως ε, έντιμοι διαμεσολαβητές και να επιδιώξουμε τα στρα... τις στρατηγικές προτεραιότητες του ευρωπαϊκού μας προγράμματος σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ε, πάρα πολύ σημαντική παρουσίαση. Τώρα περνάμε στο γύρο των ερωτήσεων και απαντήσεων. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο πρώτος, η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που είστε εδώ σήμερα. Είναι χαρά μας να συνεργαστούμε με την ε, Μαλτέσκη Προεδρία και εξεπλάγει από τις εθνικές αλλαγές που κάνατε στην ομοθεσία σας για το διαζύγιο και αντίστοιχα ζητήματα. Φαίνεται ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία στη χώρα σας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ε, διαπίστωσα ότι αναφερθήκατε και στην νομοθετική πρόταση για τις διαδικτυακές πωλήσει ε, υλικών αγαθών. Και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκαναν αυτό το λεγόμενο refit που το αποκαλούν ε, τον περασμένο Σεπτέμβριο και ξαφνικά από αυτό το refit ε, με το μαγικό ραβδάκι προέκυψε μια πολύ μεγάλη επέκταση του πεδίου εφαρμογής όχι μόνο για τις διαδικτυακές αλλά και τις εκτός δικτύου πωλήσει. Και όπως ε, καταλαβαίνετε δεν γνωρίζω τίποτα αυτή τη στιγμή που να επηρεάζει τόσο πολύ τα δικαιώματα του οποιονδήποτε, του οποιοδήποτε, είτε είναι ε, καταναλωτές είτε πολιτές. Ε, αυτό που με απασχολεί λοιπόν είναι κατά πόσο θεωρείτε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα μετά από αυτή την επέκταση και ε, ξέρω ότι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, χάρηκε και πάρα πολύ με την ιδέα να συνεχίσει την αξιολόγηση αντικτύπου και τώρα την ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάνει αξιολόγηση αντικτύπου της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής. Θα ήθελα επίσης να μας περιγράψετε λίγο και την διάθεση και τις κινήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο, διότι ξέρω ότι η κατάσταση είχε παραλύσει στο Συμβούλιο. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η διαδικασία γιατί άπτεται πάρα πολλών δικαιωμάτων και αν πραγματικά θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αρμονισμένο περιβάλλον τότε ε, μπορεί να καταλήξουμε ε, σε μια κατάσταση που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να αποφύγουμε, να περιορίσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών σε κάποιες χώρες. Ευχαριστώ. Κυρία Χάουταλα, ο κύριος ε, Ζιέφκα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό για την παρουσίαση και την πολύ ακριβή ε, περιγραφή των περιορισμών προτεραιοτήτων της Μαλτέζικης Προεδρίας του επόμενου εξαμήνου. Και ε, χαιρόμαστε γιατί το πρόγραμμα δεν είναι υπερβολικά φορτωμένο και πλούσιο που θα ήταν δύσκολο να το υλοποιήσει οποιοδήποτε. Λίγα και ε, συγκεκριμένα πράγματα που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε με στενή συνεργασία ε, του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και με τις προηγούμενες Προεδρίες. Συγχαρητήρια λοιπόν. Εγώ ε, είμαι ο εισηγητής για την αναθεώρηση του κανονισμού των Βρυξελών 2α. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα. Ο κανονισμός αυτός, ε, Βρυξέλλες 2α, όπως σωστά είπατε, και χαίρομαι που είπατε ότι είναι ιδιαίτερα προσφυλής ε, σε εσά ο κανονισμός αυτός ε, για τις Βρυξέλλες 2α, ε, γιατί αφορά πολύ σημαντικά θέματα, οικογενειακά ζητήματα που σε μεγάλο βαθμό αναπόκεινται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών αλλά υπάρχουν κάποιοι τομείς που εμπίπτουν στην κοινοτική αρμοδιότητα και είναι περιορισμένοι. Και εδώ έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ουσιαστικά ασκεί ένα συμβουλευτικό ρόλο περισσότερο αλλά ακόμη και αυτό, ο συμβουλευτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σημαντικός για τα οικογενειακά ζητήματα. Και νομίζω ότι η κοινή μα υποχρέωση και κοινό μα καθήκον είναι το εξή. Η αναθεώρηση του κανονισμού των Βρυξελών 2α για θέματα που ε, θα επιληθούν σε κοινοτικό επίπεδο θα να διευκολύνουν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών, ακόμη και για τα οικογενειακά ζητήματα και ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τη μεγαλύτερη κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών, την αλλαγή του τόπου διαμονής ή την αλλαγή του τόπου κατοικίας. Ε, δεν πρόκειται να σας ασκήσουμε πίεση για να επισπεύσετε τις εργασίες. Γι' αυτό καλύτερα να μην βιαστούμε, αλλά να σπεύσουμε βραδέως για να έχουμε και θετικά αποτελέσματα. Θα θέλαμε όμως να δούμε ποιο είναι το κλίμα στο Συμβούλιο. Ποια είναι η γνώμη του Συμβουλίου για αυτά τα σημαντικά θέματα σε σχέση με τον, την αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 2α. Έχει ήδη προσδιοριστεί κάποιο χρονοδιάγραμμα μας αναφέρατε κάποιο χρονικό ορίζοντα, αλλά είναι αρκετά απομακρυσμένος. Υπάρχει κάποιο προκαθορισμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες και τις συζητήσεις που ξεκινήσαμε για το θέμα αυτό με τη Σλοβακική Προεδρία. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Σιέφκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για τις εξηγήσεις σας και για την παρουσίασή σας. Είπατε ότι είναι ευαίσθητη η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν γέννη και της Επιτροπής μας πιο συγκεκριμένα για κάποια θέματα τα οποία σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και μας ιδιαίτερα εδώ στην Επιτροπή, διότι υπήρξε αντικείμενο και εδώ ε, στην Επιτροπή ψηφίσαμε και ψηφίσαμε και στην Ολομέλεια για την ε, φοροδιαφυγή και τις αναφορές αναχώρα ε, και για την Επιτροπή και, την, ε, και για το, ΛΟΜΕ, το Κοινοβούλιο εν γέννη είναι μια πολύ σημαντική πρόοδος. Ξέρετε κύριε Υπουργέ, εμείς ε, στο Συμβούλιο γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων νομικής φύσεως. Θα σας μιλήσω από νομικό σε νομικό. Πρόκειται για τη νομική βάση. Το θέμα της νομικής βάσης αφήνω στην άκρη την ουσία Βέβαια δεν είναι θέμα ανούσιο η ε, νομική βάση. Ξέρετε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θεωρούν ότι πρόκειται για συνήθη διαδικασία ε, της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Συμβούλιο φαίνεται να θεωρεί και νομίζω ότι αυτή ήταν η θέση που υιοθέτησε και η Μάλτα. Ε, θεωρούν λοιπόν ότι ε, πρέπει να υπάρχει ομοφωνία για το θέμα αυτό. Επομένως, ε, θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον αυτή είναι η θέση που θα υιοθετήσει και η Μαλτέρικη Προεδρία και αν αυτό το σχέδιο οδηγίας ε, προχωρήσει θα βρεθεί στάσιμο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας ή θα δεχτείτε να εργαστείτε με πιο επικοδομητικό πνεύμα. Ευχαριστώ κύριε Ντουρά. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Θα ήθελα να εκφράσω κάποιες σκέψεις πρωτού δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου που είναι μαζί μου. Να πω λοιπόν κάποια πράγματα Κυρία Χάουταλα, σας ευχαριστώ πολύ για τον τρόπο με τον οποίο μιλήσατε για το συνολικό πακέτο για τις επιγραμμικές πωλήσει. Φυσικά, το ζήτημα της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής ε, είναι ένα ζήτημα γύρω από το οποίο υπήρξαν πολύ έντονες συζητήσεις. Με ρωτήσατε αν, αν είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να το επιλύσουμε το θέμα που έχει ανακύψει. Πρέπει να σας πω ότι όχι. Βέβαιος δεν μπορώ να είμαι ότι θα καταλήξουμε σίγουρα σε κάποια λύση. Παρ' όλα αυτά δουλεύουμε στο θέμα αυτό. Οι εμπειρογνώμονές μας ε, καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες και θα δούμε τι θα γίνει. Ε, αναφέρθηκε και ο κανονισμός ε, Δουβλίνο 2α από τον κύριο Σιέφκα. Συμφωνώ on 2 2α. Ε, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ και ε, μας ενδιαφέρουν πολύ και τα σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ομοφύλων ε, και ευρύτερα τα δικαιώματα της ΛΟΑΔ κοινότητας. Είναι ένα ζήτημα που αξίζει να συζητηθεί ε, αν και δεν είμαι σήμερα αυτή τη στιγμή για να σας πω τις προσωπικές μου απόψεις ε, εκπροσωπώ το Συμβούλιο και το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δικασία ε, χάραξης των κόκκινων γραμμών της πάντως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Βρυξέλλες 2α είναι ένα ε, ένας κανονισμός πολύ σημαντικός για ε, μας γιατί ακριβώς βρίσκεται στην καρδιά των, της ζωής των ανθρώπων γιατί ε, ε, ε, μπορεί κανείς να, μεταφέρει, να μεταφέρει τα, τη ζωή του στην ουσία σε μια άλλη χώρα χωρίς να αντιμετωπίσει τεράστια γραφειοκρατικά εμπόδια. Και αυτό ήταν άλλωστε και η ουσία του ευρωπαϊκού εγχειρήματο από την αρχή. Όσον αφορά τις ερωτήσεις του κυρίου Τζουλόν, θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου για να ε, απαντήσει με περισσότερες λεπτομέρειες. Ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, ο κύριος Καουντόνα έχει την, ε, την χαρά και την τιμή να απαντήσει στον κύριο Τον. Να είναι εύκολη η ερώτηση που μου έθεσε ο Πασκάλ. Προτού όμως ε, απαντήσω στο ερώτημα του Πασκάλ, θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποια άλλα ε, στοιχεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι ε, η δική σας επιτροπή είναι ε, η πρώτη επιτροπή στην οποία εμφανίζομαι, θα παραστώ ως πρόεδρος του Συμβουλίου και αυτό σηματοδοτεί και την επιθυμία μας να υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ της Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και δεν είναι μόνο η παρουσία μας εδώ σήμερα, αλλά και το γεγονός ότι σημειώνουμε και καταγράφουμε ε, αυτά που αναφέρονται από τους συμβουλευτές της Επιτροπές και προσπαθούμε, ε, χρησιμοποιούμε όλα όσα λέγονται, ε, να τα αξιοποιήσουμε, να εξεύουμε συμβιβασμούς μεταξύ των διαφορετικών απόψεων που εκφράζονται και αυτήν την οδό θα ακολουθήσουμε και τους επόμενους έξι μήνες. Να μπω τώρα σε κάποια πιο συγκεκριμένα ζητήματα και στη συνέχεια θα ολοκληρώσω με την ερώτηση του Πασκάλ. Η Προεδρία μας κατανοεί την σημασία του ε, Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου. Αποτελεί ε, ένα στοιχείο ε, κεντρικό της ευρωπαϊκής φυσιογνωμίας και υπάρχουν και δύο σχετικές προτάσεις. Πρώτον είναι ο κανονισμός για τη φορητότητα. Εμείς ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ να προχωρήσουμε το φάκελο αυτό από εκεί που τον αφήσαμε μετά τον πρώτο τριμερή διάλογο και πιστεύουμε πραγματικά ακράδαντα ότι μπορούμε να βρούμε ε, έναν επικοδομητικό συμβιβασμό προκειμένου να καταλήξουμε, να σε μια πρώτη συμφωνία στη διάρκεια της δικής μας Προεδρίας. Στην διάρκεια λοιπόν, ε, στον τομέα αυτό όσον αφορά τα, πνευματικά δικαιώματα, την ε, συνθήκη του Μαρακές, πρέπει να σας πω ότι πιστεύουμε στη σημασία της ε, συνθήκης αυτής και, την, και, στη, και, στη μοναδική ευκαιρία που παρέχει στους ε, αμβλίωπες ανθρώπους και γι' αυτό ε, ελπίζουμε να καταφέρουμε να κυρώσουμε την συνθήκη αυτή μόλις αποφανθεί το δικαστήριο όσον αφορά τις αρμοδιότητες η Κομισιόν τον τελευταίο Σεπτέμβριο εξέδωσε δύο εκτελεστικούς κανονισμούς όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της συνθήκης και ελπίζουμε ότι αυτό θα μας βοηθήσει προκειμένου να ε, προσαρμόσουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο στις απαιτήσεις αυτής της συνθήκης. Και δεδομένης της πολιτικής βούλησης και των δύο συνομοθετών ε, να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το έργο αυτό δηλαδή εντός της Μαλτέζικης Προεδρίας. Ε, θα υπάρξουν βεβαίως και συζητήσεις και στη δική σας επιτροπή ε, και αναμένουμε και την έκθεση του κύριου Μαξ Άντερσον και περιμένουμε τους επόμενους μήνες να εγκριθεί και η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Η Προεδρία θα εξακολουθήσει να εργάζεται επί της πρότασης της Κομισιόν για την, τον εξυγχρονισμό του συστήματος πνευματικών δικαιωμάτων στη νέα ψηφιακή εποχή στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Ο κύριος στόχος μας θα είναι να εξασφαλίσουμε την σωστή ισορροπία μεταξύ της ελεύθερης ε, κυκλοφορίας πληροφοριών, της διατήρησης ε, της ε, πολιτικής κληρονομιάς από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά τα δικαιώματα των δημιουργών και του περιεχομένου. Και στις συζητήσεις που γίνονται στο Συμβούλιο Έχουμε δεσμευτεί να σημειώσουμε όσο μεγαλύτερη πρόοδο γίνεται. Έχουμε ξεκινήσει ήδη με μια ανταλλαγή απόψεων. Ε, ε, έχετε ξεκινήσει μάλλον ήδη μια ανταλλαγή απόψεων εδώ στην Επιτροπή Γιούρη ε, για την οδηγία για τα, για πνευματικά δικαιώματα όπου η κυρία Κομοντίνη είναι η συγγήτρια και προσβλέπουμε στην δική της συνεργασία και στις εξελίξεις από εδώ και πέρα και με επικεφαλή στον Τίτμαρ Κέσνερ. Όσον αφορά τις ε, εκθέσεις αναχώρα και την ε, βελτίωση της νομοθεσίας. Ε, μιλήστε λέει, λέει η Πρόεδρος, αλλά μην ξεχάσετε να απαντήσετε και στον κύριο Τζιρόν. Μα προσπαθώ να κερδίσω χρόνο και Όσον αφορά την, ε, το ζήτημα της βελτίωσης νομοθεσία, εμεί θα συνεχίσουμε τι προσπάθειε μα για την εφαρμογή της Διοργανικής Συμφωνίας για την καλύτερη νομοθεσία, που συνυπογράφηκε από τα τρία θεσμικά όργανα τον Απρίλιο και η συμφωνία αυτή αποσκοπεί στο να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθετεί προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλή ποιότητα της νομοθεσίας και να εξασφαλίζεται ότι η νομοθεσία αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Συλλογικά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να θα εργαστούμε για την ε, λήψη μέτρων ε, και την θέση θέσπιση νομοθεσίας που θα βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και που θα άρει ε, παλαιά εμπόδια γραφειοκρατικά. Ε, αυτό θεωρούμε ότι είναι και η ουσία της Διοργανικής Συμφωνίας για την καλύτερη νομοθεσία από την άποψη της συγκρισιμότητας ε, θα εξετάσουμε την, ε, το πρόγραμμα REFIT της Κομισιόν και θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε και εμείς από την δική μας πλευρά για τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος ε, και κλίματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις ευρύτερα. Θα προσπαθήσουμε επίσης να εργαστούμε στη βάση της ανακοίνωσης της Κομισιόν που δημοσιεύτηκε πρόσφατα και θα ε, διενεργήσουμε και μελέτες αντικτύπου ε, όσον αφορά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις προκειμένου η νομοθεσία που θα θεσπίζεται από εδώ και πέρα να έχει απτά θετικά αποτελέσματα στη ζωή των ε, πολιτών μας. Τέλος, θα προσπαθήσουμε να άρουμε κανονιστικά εμπόδια για την καινοτομία ε, κάτι που είναι κρίσιμη σημασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά, ε, πολιτικά και ε, περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει λοιπόν η έρευνα να γίνει πιο καινοτόμα και θα προσπαθήσουμε σε αυτόν τον τομέα να σημειώσουμε πρόοδο ακριβώς γιατί ο τομέας αυτός επηρεάζει, έχει άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων και στις αλλαγές που έχουν επισυμβεί στις ζωές των ανθρώπων το, τα τελευταία χρόνια για να προσπαθήσουμε να αποσβέσουμε τους κραδασμούς των αλλαγών αυτούς. Ε, θα υπάρξουν λοιπόν συζητήσεις, διαβουλεύσεις μεταξύ εμπλεκομένων φορέων, κρατών μελών, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το CBCR. Ε, στον τομέα αυτό και στο θέμα αυτό τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να εξετάζουν τη νομική βάση της, νομικής, ε, της πρότασης κομισιών. Ε, περιμένουμε ακόμη αυτήν την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας και την ε, γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου Παρ' όλα αυτά μπορούμε ήδη από τώρα να βασιστούμε στο πολύ θετικό έργο που επιτέλεσαν η Ολλανδική και η Σλοβακική Προεδρία. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου λοιπόν εμείς προσβλέπουμε, να, προβλέπουμε μάλλον να σημειώσουμε σημαντική προοδό το επόμενο διάστημα και ε, επιδιώκουμε να σημειώσουμε πρόοδο και στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, ανάμεσα στα κράτη-μέλη, την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Thank you, Minister. ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κυρία Κομοντίνη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους δύο υπουργούς που εκπροσωπούν τη Μαλτέζικη Προεδρία. Ο Υπουργός ε, Καρδόνα ε, μας υπονόησε ότι ε, οι συζητήσεις για το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων έχουν ξεκινήσει ήδη στο Συμβούλιο. Ως που είμαι αρμόδια για το θέμα αυτό, ε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είναι αμφολεγόμενη η φύση αυτού του θέματος ε, και είναι πολύ περίπλοκη συζήτηση που διεξάγεται και εντό του Κοινοβουλίου αλλά και με τους ενδιαφερομένους και από τους ενδιαφερομένους. Εσείς όμως είπατε ότι οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει και στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μας πείτε ποια θέματα από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δημιουργούν ε, τις περισσότερες ε, διαμάχες ε, στο Συμβούλιο και ποιες πλευρές της Πρώτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρείτε εσείς προτεραιότητα. Ευχαριστώ Τερέζη, κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω και τους δύο υπουργούς που ε, μας έκαναν την παρουσίασή τους. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε για τη συνθήκη του Μαρακές, αλλά και αυτά που είπατε και εσείς κύριε Μπονίτσι, όσον αφορά τις προσπάθειες για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Όλα αυτά είναι πολύ καλά νέα. Ε, θα ήθελα να επιμείνω σε ερωτήσεις για τις ε, εκθέσεις αναχώρα για την ε, φορολογική βάση. Σας ευχαριστούμε που μας δώσετε αυτές τις συνολικές εξηγήσεις ε, για την ερώτηση του συναδέλφου και θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί. Αυτό το οποίο βλέπουμε μέχρι τούδε από αυτά που κάνει το Συμβούλιο και τις εργασίες οι οποίες έγιναν στη διάρκεια της Σλοβακικής Προεδρίας πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι είναι αρκετά ζωφερό. Ε, δεν αναφέρομαι μόνο στη νομική ερμηνεία που δίνει το Συμβούλιο, που εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπουμε με εντελώ διαφορετικό τρόπο και είμαι και πεπισμένη ότι έχουμε δίκιο, αλλά αναφέρομαι και στις διαπραγματεύσεις μέχρι τώρα όσον αφορά το περιεχόμενο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω προς ποια κατεύθυνση θα μπορούσατε να κινηθείτε όταν συζητούμε αυτά τα οποία ε, συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στις ομάδες εργασίας στο Συμβούλιο για τη συμμόρφωση και να εξηγήσετε. Αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε η όλη πρόταση να κατευθυνθεί ε, και προς άλλη κατεύθυνση, διότι ε, πάμε πλέον στο παράλογο και τα κράτη-μέλη φαίνεται ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν με πρόσχημα τη νομική βάση έναν τρόπο να ξεφύγουν. Ε, θα ήθελα να ξέρω την προπτική, την εικόνα που έχετε εσείς αυτή τη στιγμή ε, για ε, το θέμα αυτό και προς ποια κατεύθυνση θα μπορούσε να κινηθεί. Σήμερα το πρωί, ε, δεν θα ήθελα να επισέλθω σε λεπτομέρειες, στη που κάναμε και κλεισμένο των ε, είχαμε μια παρουσίαση και ακούσαμε και το Συμβούλιο για την νομική βάση και έμεινα με την εντύπωση ότι το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή δεν είναι διατημένο να προχωρήσει και να χρησιμοποιήσει όλη αυτή την ορμή που έχει προκύψει από το θέμα. Όταν παρουσιάστηκε ε, η πρόταση του Επιτρέπου Χιλ ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα πράγματα γιατί αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι αποδυναμημένο το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, Εύελιν. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να θέλει να ε, πάρει το λόγο. Κύριε Υπουργέ. για να απαντήσω σε αυτό που είπε η Τερέζα. Το Συμβούλιο έχει ξεκινήσει ε, τις συζητήσεις και θα συνεχίσουμε. Ε, είναι θέμα προτεραιότητας για τη Μαλτέζικη Προεδρία την εξέταση των δύο προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στόχο έχουν να εξυγχρονίσουν την, ε, το επιχειρηματικό νομικό πλαίσιο στο ψηφιακό περιβάλλον. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν αναλυτικά και ο βασικός μας στόχος ω Συμβούλιο είναι να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε την κατάλληλη ισορροπία ε, αφενός, όπως είπα προηγουμένως, ε, για την ελεύθερη ροή πληροφοριών, την δημοσιοποίηση και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και αφετέρου τα δικαιώματα του δημιουργού του περιεχομένου. Και αυτά είναι θέματα τα οποία εξετάζουμε προκειμένου να ε, έχουμε και έναν επικοδομητικό διάλογο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή θα έχουμε προχωρήσει αρκετά και στα δύο όργανα. Προφανώς είμαστε σε πλήρη ταχύτητα, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Τίνουμε δίκονου σε αυτά τα οποία λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά όταν θα καταλήξουμε και στα εσωτερικά μας συμπεράσματα θα προχωρήσουμε. Σκοπεύουμε επίσης να προχωρήσουμε και τις συζητήσεις που όπως σας είπα στην εισαγωγή μου ε, Μα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, είναι μεγάλη προτεραιότητα, ιδιαίτερα στα πλαίσια τη συνθήκη του Μαρακέ. Ήταν προτεραιότητα και στη Σλοβακική Προεδρία και όταν αντιμετωπιστούν και οι εκκρεμότητες που υπάρχουν σε τεχνικό επίπεδο και συζητήσουμε και με τους ενδιαφερομένους, είμαστε βέβαιοι ότι θα καταλήξουμε σε ένα υγιές επίπεδο ώστε να έχουμε και συμφωνία στη διάρκεια της Προεδρίας μας. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, που αφορά και πάλι τις εκθέσεις αναχώρα. Νομίζω ότι είναι λίγο πρόημο αυτή τη στιγμή να κάνουμε εικασίες για το προς τα ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Είναι κάτι βεβαίως που είναι πολύ λεπτό για τα κρατη και η Προεδρία μας είναι πεπισμένη ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για την καταπολέμηση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης. Έχουμε λοιπόν μια επικοδομητική στάση και ε, είναι και η στάση των αντιπροσωπιών σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και θέλουμε να συνεχίσουμε από την καλή πρόοδο ε, στην οποία κατέληξαν οι προκάτοχοί μας, ε, οι κάτω χώρες και η Σλοβακία. Ο στόχος ε, βεβαίως είναι να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το, Συμβούλιο, με το Κοινοβούλιο ε, και πιθανή συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Αυτή τη στιγμή θα προχωρήσει και το Συμβούλιο τις εσωτερικές του διαδικασίες και θα ολοκληρώσει και τις εκθέσεις του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου και πάλι, όπως σας είπα προηγουμένως, έχει γνωμοδοτήσει επί του θέματος. Αυτό θα οδηγήσει σε μια ειδική νομοθετική διαδικασία με ομοφωνία στο Συμβούλιο και διαβούλευση ε, με το Κοινοβούλιο. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι αντίθετη σε αυτή την αξιολόγηση. Δεν υπάρχει ομοφωνία στο Συμβούλιο για την αλλαγή της νομικής βάσης και οι συζητήσεις συνεχίζονται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλο, άλλος κανείς να θέλει το λόγο. Οπότε δεν μου μένει παρά να ευχαριστήσω θερμά τους δύο υπουργού για την παρουσία τους και την παρουσίαση που μας έκαναν των προτεραιοτήτων τους. Και κρίνοντας από τις απαντήσεις, ε, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και πολύ εύκολο το έργο σας. Σας εύχομαι λοιπόν καλό κουράγιο, ενέργεια και καλή επιτυχία μαζί με την απαραίτητη τύχη που θα χρειαστεί η Μαλτέζικη Προεδρία. Ευχαριστώ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, may I ask to, σας παρακαλώ λίγη ησυχία για να συνεχίσουμε. Παρακαλώ, καθίστε. Περνάμε στο επόμενο σημείο της της διάταξης και θα δώσω το λόγο στον κύριο Σβιεύκα. Παρακαλώ. Και σας ε, θέρμα παρακαλώ λίγη ησυχία. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Εκπροσωπώ εδώ τον ε, πρόεδρό μας, τον κύριο Σφόποντα, που απουσιάζει γιατί έπρεπε κατεπηγόντως να επιστρέψει στην Πράγα. Για να μην ε, χάσουμε χρόνο όμως, με παρακάλεσε να, τον παρουσια... να παρουσιάσω εγώ την ε, γνωμοδότησή του. Τη γνωμοδότηση που πραγματεύεται το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δεν πρόκειται για ένα καινούριο θέμα, δεν είναι πρωτοφανές, το έχουμε ήδη εξετάσει. Συζητήσαμε τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει και ο πρόεδρος Σβόμποντα στην γνωμοδότησή του, που είναι πολύ συμπυκνωμένη και πολύ μεστή, προσπάθησε να επικεντρωθεί σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος γιατί τα σημαντικότερα στοιχεία της γνωμοδότησης αφορούν τη λειτουργία της δικτυακής, διαδικτυακής πύλης της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης. Θεωρεί ο κύριος Παμπότα την πύλη αυτή σημαντικό εργαλείο για την πρόσβαση σε πληροφορίες στη δικαιοσύνη και όλο και περισσότεροι πολίτες χρησιμοποιούν αυτή τη δικτυακή πύλη. Ε, η ανάπτυξη λοιπόν ε, τέτοιων ε, ψηφιακών εργολείων είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορούν οι πολίτες γρήγορα, με ακρίβεια και αποτελεσματικά να ενημερωθούν για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Ε, τέτοιες προτάσεις εξυπηρετούν και τις επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν και πολλές πτωχευτικές διαδικασίες και τα μητρώα οπότε ένα τέτοιο, μια τέτοια προσπάθεια για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών συναλλαγών εξυπηρετεί όχι μόνο τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις. Ο εισηγητής σας παρακαλεί να λάβετε υπόψη την προσέγγιση του κατά την εκπόνηση της γνωμοδότησης. Εσκεμένα επικεντρώθηκε σε ζητήματα αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Γιούρη. Οπότε και εσείς, κατά τη σύνταξη των τροπολογιών σας, περιοριστείτε, παράκληση του εισηγητού, ε, παρακαλείστε να περιοριστείτε σε τέτοιου είδου θέματα, στι δικέ μας αρμοδιότητες. Έτσι θα γίνει πιο συνεκτική η γνωμοδότηση, αλλά θα είναι και πιο αποτελεσματικό το έργο μας. Ε, 10 ή μάλλον όχι, 16, 16 Ιανουαρίου λίγη προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών έχουν μείνει ακόμη λίγες μέρες δηλαδή για να εκπονήσετε και να καταθέσετε τις τροπολογίες σας. Αυτά κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς κύριε Σεβιεύκα. Θέλει κανείς παρακαλώ το λόγο μετά την ενημέρωση που μας έκανε ο κύριος Βιεύκα. Δεν βλέπω κανένα θελοντή. Οπότε μπορούμε να περάσουμε ήδη στο επόμενο σημείο της ημερήσης διάταξης. που είναι το σημείο 23 Το σημείο 23 λοιπόν του κυρίου Ζήλε Μπρετών. Merci, euh, euh, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησής μου για την απαλλαγή του 2015 Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το σχέδιο γνωμοδότησης είχα ήδη την ευκαιρία να σας το υποβάλω. Κατατέθηκα γι' αυτό 13 τροπολογίες, τις οποίες θα ήθελα συντομία να σχολιάσω. Επί των 13 τροπολογιών, τέσσερις από αυτές επιχειρούν να τροποποιήσουν ε, ένα εδάφιο που είχα συντάξει και που ίσως θέλει λίγο εκτός θέματος γιατί έλεγε ότι δεν ήταν απαραίτητη η μεταρρύθμιση του δικαστηρίου γιατί εγώ σχολίαζα κάποια στοιχεία που έδειχναν πόσο ικανοποιητική είναι η δραστηριότητα του δικαστηρίου και είπα ότι κατά τη γνώμη μου επιβεβαιώνεται ότι η μεταρρύθμιση του δικαστηρίου δεν είναι απαραίτητη. Άλλωστε δεν ήταν μυστικό ότι εγώ ήμουν κατά της μεταρρύθμισης. Γι' αυτό και οι συνάδελφοι κατέθεσαν τέσσερις τροπολογίες οταν τη διαγραφή αυτού του σημείου. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει συνένεση υπέρ της διαγραφής αυτού του στοιχείου. Οι ε, τροπολογίες 1 και 4 μιλούν για το θέμα αυτό. Η κυρία Χάουταλα αντίθετα πιστεύει ότι ακριβώς τα στοιχεία που έδωσα καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης. Οπότε καλύτερα να διαγράψουμε αυτό το εδάφιο όπως προτείνουν οι τροπολογίες 2, 3 και 4. Χρυσόγονος, Καβαντά και Μπούντα ήταν οι συντάκτες των τριών τροπολογιών. Νομίζω η πιο λογική τροπολογία είναι αυτή του κυρίου Καβαντά, που απλώς ζητά διαγραφή ε, της ε, φράσης που περιείχε το σχόλιο για τη μεταρρύθμιση του δικαστηρίου και δεν τροποποιεί την τεχνική ε, σχετικά περιγραφή που γινόταν παραπάνω. Οι άλλες δύο τροπολογίες Χρυσόγονο και Μπούντα λίγο τροποποιούσαν τη διατύπωση. Δεν νομίζω όμως ότι ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικέ οι τροπολογίες τους, γιατί ε, εκεί που λέγω ικανοποιητικό επίπεδο δραστηριοτήτων προτείνεται να βγει ιδιαίτερο επικοδομητικό. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ επικοδομητικό γιατί ναι, με θαυμάζουμε το δικαστήριο, αλλά δεν είναι και τέλεια τα πράγματα, έχονται βελτιώσει. Και αν πούμε ιδιαίτερω ικανοποιητική ή πολύ ικανοποιητική δραστηριότητα του δικαστηρίου, μα στερεί τη δυνατότητα να ζητήσουμε στη συνέχεια βελτιώσει. Αυτά και από τι τέσσερι τροπολογίε που ζητούν διαγραφή, ε, εγώ είμαι υπέρ τη τρία. Μετά έχουμε διάφορες τροπολογίες για διάφορα θέματα. Η τροπολογία 5 ζητά προσθήκη νέας πρωτοβουλίας που εθαρρύνει τη λήψη ε, μέτρων ε, και ναυσμάτων για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα των δικαστών. Αυτό το πνεύμα της γνωμοδότησης, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να γυρίζουμε το μαχαίρι στην πληγή εδώ. Γιατί μερικές φορές ε, το καλύτερο είναι ο του καλού. Δεν θα πρέπει να αναγάγουμε ως αυτό σκοπό την παραγωγικότητα των δικαστών. Γιατί το θέμα είναι να αποδίδεται με νυφάλιο τρόπο η δικαιοσύνη και να είμαστε και λογικοί στι απαιτήσει μα. Νομίζω ότι η παράγραφο αυτή είναι κάπω ανησυχητική η σχετική τροπολογία. Είμαι λοιπόν κατά τη τροπολογία 5 του κ. Χρυσόγωνου. Τροπολογία 6 τώρα του κ. Μπούντα. Παρά είναι ενθουσιώδη. Ναι, με τα στοιχεία που δίνω για την παραγωγικότητα του δικαστηρίου είναι θετικά, αλλά το να λέμε ότι η αιτήσια ε, δραστηριότητα ε, φτάνει σε ένα πρωτοφανές ε, επίπεδο άνευ προηγουμένου στην ιστορία του δικαστηρίου, νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Γιατί έτσι αποδυναμώνουμε τα υπόλοιπα μας σχόλια. Τροπολογία 7 του κυρίου Μπούντα και πάλι. Ε, αρκετά ενδιαφέρουσα η τροπολογία αυτή. Προτείνει την προσθήκη μιας παραγράφου που ουσιαστικά δίνει ένα νέο στοιχείο που είχα παραλείψει εγώ που είναι αρκετά ενδιαφέρον. Σας το διαβάζω λοιπόν. Στην παράγραφο αυτή ε, εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας γιατί οι ε, υποθέσεις που έχουν διαθετηθεί ε, αυξάνονται κατά 5 7, από 5 σε 7%. Είναι πολύ θετικό και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Γι' αυτό και με υπέρ της τροπολογίας 7. Η τροπολογία 8 του κυρίου Μπούντα τώρα είμαι κατά, γιατί κάνει μια αξιολογική κρίση για τη μεταρρύθμιση του, δικαστηρίου. Ε, μια και όμως προκάλεσε κατακραυγή αυτή η ατυχής μου πρόταση, εγώ θα έλεγα να αφήσουμε κατά μέρος το θέμα της μεταρρύθμισης του δικαστηρίου. Δεν είναι της παρούσης απαλλαγής. Τροπολογία 9, του κυρίου Μπούντα και πάλι. Αρκετά μακροσκελής και αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία άσκησης ε, προσφυγής προς το δικαστήριο. Εγώ περιλαμβάνω μία σύντομη παραγραφό. Ο κύριος Μπούντα διπλασιάζει το εύρος της παραγράφου. Δεν πολύ συμφωνώ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κιόλα. Γιατί ενθαρρύνουμε κα... κατά συνέπεια τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα για να προωθήσουν τη χρήση αυτής της εφαρμογής και ούτω καθεξής. Αλλά δεν είμαι πεπισμένο για την αναγκαιότητα αυτή τη τροπολογία. Τροπολογία 10, στο ίδιο πνεύμα και αυτή, προσπαθεί να αναπτύξει την παραγραφό, να την εμπλουτίσει. Δεν συμφωνώ. Λέει απλώς ότι η ηλεκτρονική υποβολή επιτροπεί την ε, ηλεκτρονική ανταλλαγή των δικογράφων. Νομίζω ότι αυτό είναι προφανές, δεν χρειάζεται να το ε, επισημαίνουμε. Και τώρα χρειάζεται μια τροποποίηση της παραγράφου 6, γιατί και αυτή η παράγραφος ε, έδωσε λαβή για τροπολογίες. Εγώ θα πρότεινα την τροπολογία 11 του κυρίου Χρυσόγονου, που έχει δύο πλονεκτήματα σε σχέση με τη δική μου πρόταση. Καταρχήν διορθώνει το ύφο της δικιάς μου παραγράφου, γιατί ε, η δικιά μου παράγραφος 6 δεν ήταν και πολύ σωστή. Οπότε αντί να λέμε όπως έχει αποδείξει, να πούμε ε, όπως έχει αποδειχθεί, να πούμε όπως έχει αποδείξει. Επίσης προτείνει τη συμπερίληψη μιας σύντομης παραγράφου που είναι ενδιαφέρουσα από δημοκρατικής πλευράς. Επιμένει στην ανάγκη να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες ως προς την ύπαρξη αυτής της εφαρμογής και των πλεονεκτημάτων της. Καλό να υπενθυμίζουμε ότι η ηλεκτρονική διαδικασία έγινε χάρη του κοινού. Γι' αυτό και θα πρέπει να ενημερωθεί το κοινό γι' αυτό. Ενδιαφέρον λοιπόν αυτό. Και οι δύο τελευταίες τροπολογίες, τροπολογία 12 τη κύρια Χάουταλα, δεν θα έλεγα ότι είναι περίτη άχρηστη, αλλά μιλά για την ισότητα. Αυτό όμω το έχουμε αναφέρει αλλού. Εγώ ε, είχα ω ε, ζητούμενο την ισότητα ανδρών και, και γυναικών. Τώρα να προσθέσουμε σε αυτό το θέμα της ισορροπίας ανδρών και γυναικών ένα κεφάλαιο για την ισότητα, δεν το κρίνω σκόπιμο, γιατί εξετάζοντας τα αριθμητικά στοιχεία βλέπουμε ότι σε μερικές διοικητικές θέσεις ε, οι γυναίκες είναι η πλειοψηφία. Οπότε δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα υποεκπροσώπησης ενός φίλου στη σύνθεση του δικαστηρίου. Θα προτιμούσα λοιπόν να παραμείνουμε στη δική μου ε, διατύπωση για την ισορροπία των δύο φίλων, που είναι σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα. Και τέλος, ε, τροπολογία 13 του κυρίου Μπούντα, Ούτε και αυτή τη θεωρώ ιδιαίτερα απαραίτητη, γιατί προτείνει στην ίδια παράγραφο την προσθήκη δύο προτάσεων που τονίζουν ότι οι γυναίκε είναι το 60% του προσωπικού του δικαστηρίου. Το πρόβλημα είναι ότι ε, η παράγραφος αυτή αφορά τις ε, διευθυντικές θέσεις. Αν προσθέσουμε λοιπόν μια φράση που δεν αφορά αυτές τις θέσεις, είναι σαν να δημιουργούμε μια σύγχυση για το περιεχόμενο της παραγράφου. Αυτά και ευχαριστώ τους συναδέλφους που εκπώνησαν 13 τροπολογίες. Δεν περίμενα τόσο πολλές τροπολογίες για ένα τόσο ε, σεπτό σχέδιο γνωμοδότησης. Από τις 13 αυτές τροπολογίες είμαι υπέρ των τριών που σας ενέφερα και οι υπόλοιποι στα σκόπιμες γιατί έδωσαν λαβή για συζήτηση. Κυρία Χάουταλα, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λεμπρετών για τον ενδελεχή τρόπο με τον οποίο συζητά μαζί μας τις ε, τροπολογίες. Συμφωνώ μαζί του ότι πράγματι αν δεν κινηθούμε ε, έως το σημείο που θα ήθελε εκείνος ε, θα μπορούσαμε ενδεχομένω να διαγράψουμε συνολικά την αναφορά αυτή. Εγώ παρόλα αυτά θα επιμείνω στην τροπολογία μου σύμφωνα με την οποία μπορούμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες εξορθολογισμού. Ε, το βασικό ζητούμενο για μένα είναι να επιδιώξουμε αυτή τη μεταρρύθμιση και στη συνέχεια μπορούμε να το συζητήσουμε και με τον Λεμπρετόλ. Το περιεχόμενο της δικής, μας, της δικής μου τροπολογίας της τροπολογίας 12 είναι να υπενθυμίσουμε στα όργανα την, την κοινή διακήρυξη που έκαναν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ σύντομη. Να σας την θυμίσω λοιπόν. Δεν αφορά την ισότητα των φίλων και την εξίσωση, αλλά τη σύνθεση του Γενικού Δικαστηρίου ε, σε δικαστές. Αυτό που είχαμε αποφασίσει είναι ότι θα υπάρχουν δύο δικαστές από κάθε κράτος μέλος και για να εξασφαλιστεί η ισότητα των φύλων που είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 3 της συνθήκης οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα πρέπει στο μέγιστο δυνατό βαθμό να ε, ε, προωθούν υποψήφιους για το Γενικό Δικαστήριο με βάση τις ε, διατάξεις των σχετικών ε, άρθρων και να προσπαθούν να προωθούν ε, με ισότητα τα δύο φύλλα. Αυτό δεν μπορεί απλά να γίνει υποσημείωση, γιατί υπάρχουν ήδη κράτη-μέλη τα οποία, έχουν πει, ε, δεν, τα οποία λένε δεν έχουμε ε, γυναίκες δικαστές με τα απαραίτητα προσόντα. Να τα βρουν. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συμπεριληφθεί μια τέτοια αναφορά. Ναι, καλή πρόταση άλλο μέλος της Επιτροπής που, που θα ήθελα να παρέμβει. Κύριε Λεμπρετών, θέλετε να απαντήσετε. Όχι, όχι. Περίμενα βεβαίως την αντίδραση της κυρίας Χάουταρλα γιατί είχα καταλάβει ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο το οποίο άλλωστε ξεπερνάει και την έκταση του κειμένου μου, το οποίο είναι πολύ ταπεινό. Θα το υποβάλουμε προς ψήφιση και μετά θα δούμε, γιατί όχι. Πολύ ωραία. Ε, χαίρομαι που σας ευχαριστεί η δουλειά για το θέμα αυτό, κύριε Λεμπρετό. Alors, moi, Εμένα μου αρέσει η δουλειά του νομικού και πάντα χαίρομαι όταν ασχολούμαι με το δίκαιο, ακόμα και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. donc, on Περνάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Το θέμα της κυρίας ε, Μπερζερόν για τους ευάλωτους ενήλικες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. πρόκειται για την έκθεση αυτή λοιπόν για τους ευάλωτες ενήλικες και την ε, προστασία τους. Η συγκεκριμένη πρόταση ίδιας πρωτοβουλίας αφορά άτομα άνω των 18 ετών που ε, δεν έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν ε, το άτομό τους και τα αγαθά τους. Ε, ξέρουμε όλοι ότι ο καθής από μας μπορεί να βρεθεί άμεσα ή έμεσα σε αυτή τη θέση. Ε, μπορεί αυτή η αδυναμία να προκύψει από ψυχικούς ή από φυσικούς παράγοντες, από κάποιο ατύχημα ή λόγω γύρανσης ή από εκφυλιστικές ασθένειες οι οποίες οφείλονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Υπάρχουν ε, κάποιες διάσημες ε, υποθέσεις οι οποίες κυκλοφόρησαν και στον τύπο. Υπάρχει η περίπτωση της κυρίας Μπετανκούρ η οποία βρισκόταν σε αδυναμία λόγω της ηλικίας της και υπάρχει και ε, ε, μια άλλη πολύ γνωστή περίπτωση λόγω ε, ενός ατυχήματος. Στο «πάπι Boom που ανήκω εγώ, που είναι αναλογία του Baby Boom, ανησυχούμε ιδιαίτερα για τα προβλήματα αυτά, διότι είμαστε πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι γεννηθήκαμε στη δεκαετία του 50 και σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ε, η, ηλικία μας μας οδηγεί και σε πολλές ε, εκφυλιστικές ασθένειες. Ε, θα πρέπει λοιπόν να γίνουν κάποια πράγματα σε νομικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε κάποιος ο οποίος θέλει να πάει να ζήσει σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορεί ε, και αν έχει αποκτήσει ε, περιουσία ε, λόγω γάμου για παράδειγμα να μπορεί να κρατήσει αυτά τα αγαθά και υπάρχουν προβλήματα ορισμένες φορές λόγω του γεγονότος ότι διαμένει σε άλλη χώρα και δεν είναι η χώρα καταγωγής του. Ε, ξέρετε ότι όταν κάποιος συνταξιοδοτείται προτιμάει να πάει σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ο ήλιος να λάμπει όλη ε, το χρόνο και να μην χρειάζεται να μένει στη χώρα στην οποία γεννήθηκε. Ε, και επίσης μπορεί να υπάρξει και κάποιο τροχαίο ατύχημα. Ε, στα πλαίσια του Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ γνωστή η μεικτή οι γονείς είναι από διαφορετικές χώρες, τα παιδιά γεννιούνται σε άλλη χώρα. Τι θα γίνει όταν υπάρξει μια ασθένεια ή κάποιο ατύχημα που ε, οδηγεί σε μόνιμη αναπηρία και δεν μπορεί κάποιο να φροντίσει τον εαυτό του. Τι δίκαιο επικρατεί σε αυτή την περίπτωση, ποιο μπορεί να του βοηθήσει, ποιο μπορεί να του εκπροσωπήσει, πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγή του. Υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν τα οποία ε, οφείλονται στην προσωπική τους αδυναμία αλλά και στο γεγονός ότι ζουν εκτός συνόρων. Ε, πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτά τα ευάλωτα άτομα και να προσπαθήσουν να έχουν κάποιες συγκεκριμένες σαφείς απαντήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν επαφίεται σε εμά να καθορίσουμε ένα κατάλληλο νομικό καθεστώς για αποτελεσματική προστασία λόγω της αδυναμίας αυτών των ατόμων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η Ευρώπη δεν έχει ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να στοχεύει τα αδύναμα αυτά άτομα. Οι δομές προστασίας διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών πολύ ουσιαστικά και δεν είναι και πολύ ρεαλιστικές. Δεν προβλέπουν, για παράδειγμα, ε, ενιαία παρέμβαση σε νομικό επίπεδο, σε ε, κοινοτικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε ένα ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγγνώμη, ενέκρινε ένα ψήφισμα που ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών και να αναγνωρίζει τη εκτέλεση των αποφάσεων για τους ευάλωτες ενήλικες. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν δεν έχει ακόμα υποβάλει κάποια πρόταση. Αυτή τη στιγμή σε εθνικό και ε, ε, ευρωπαϊκό επίπεδο το βασικό ε, μέσο αναφοράς για τις διασυνοριακές υποθέσεις που αφορούν τα ευάλωτα άτομα είναι η σύμβαση της Χάγης του 13 Ιανουαρίου του 2000. Πρόκειται για ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο είναι πολύ καλό αλλά μέχρι τώρα μόνο 20 χώρες το έχουν υπογράψει και 8 τις, το έχουν κυρώσει. Μεταξύ αυτών, οι δύο δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε το Μονακό ένα από αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με το δίκαιο που προστατεύει τις χώρες, ε, τα άτομα αυτά στις διάφορες χώρες, αλλά κυρίως να υπάρχει μια ενιαία μορφή εκτέλεσης των αποφάσεων, κάτι το οποίο θα διευκολύνει τη ζωή των ευάλωτων ε, ε, ενηλίκων που έχουν διασυνοριακά προβλήματα και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Προτείνω τα εξή στην έκθεσή μου. Καταρχάς, επιθυμούμε κατεπηγόντως να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση της Χάγης που καθορίζει ένα συνεκτικό, ισορροπημένο, σαφές και συγκεκριμένο νομικό σύστημα. Πέραν όμως των ωφελών που θα μπορούσαμε να έχουμε για τα κράτη-μέλη, ε, για κάποια κράτη-μέλη θα πρέπει να γίνει πλήρης μεταρρύθμιση της νομοθεσίας και το είδαμε και στη Γαλλία, διότι έγινε μια μεταρρύθμιση το 2008, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος την ημερομηνία, κάπου τότε έγινε και ε, υπάρχει πολύ σημαντικό οικονομικό κόστος. Ε, καταλαβαίνω λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν τη διάθεση να μεταρρυθμίσουν όλοι τους την νομοθεσία για να προστατεύσουν αυτούς τους ενήλικες. Και όσον αφορά τα νομοθετικά μέτρα τα οποία ε, αφορούν ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προτιμούσαμε να υπάρχει ένας κανονισμός και όχι μια οδηγία. Δεύτερον, βασικός στόχος της οδηγίας αυτής θα πρέπει να είναι να διευκολύνουμε στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αναγνώριση και εκτέλεση των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται σε ένα κράτος μέλος και να μην υπάρχει απέτηση ε, να επαναλαμβάνονται αυτές τις διαδικασίες. Αυτό είναι το βασικό. Εάν λαμβάνετε ένα μέτρο προστασίας σε μία χώρα μέλος, θα πρέπει να αναγνωρίζετε de facto στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, χωρίς να πρέπει να είναι υποχρεωμένος κάποιος να ξεκινήσει τη ε, διαδικασία εκ του μηδενός. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν πλήρη δικαιώματα για την απόφαση που ελήφθη και θα πρέπει να υπάρχουν ενιαία έντυπα για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πιστοποιούν ότι υπάρχουν μέτρα προστασίας ή κάποια εντολή ε, αδυναμίας καθώς και επίσης ένα ευρωπαϊκό έντυπο το οποίο θα υποδεικνύει τι δυνατότητες έχει το άτομο το οποίο αναλαμβάνει ε, να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα προστασίας. Ε, ο στόχος αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας είναι να βελτιώσουμε την ε, ε, επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών. Το να υπάρχει μια ενιαία αρχή όπως προβλέπει η Σύμβαση της Χάγης σε κάθε κράτος μέλος που θα ασχολείται με τα θέματα αυτά θα βοηθήσει. Αυτές οι κεντρικές αρχές ε, θα διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών καθώς επίσης και την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τους ευάλωτους αυτούς ενήλικες και ε, σε θέματα που αφορούν την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα τους. Επίσης, προκειμένου να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτές τι πληροφορίες, θα πρέπει σε κάθε κράτο μέλος να υπάρχουν μητρώα τα οποία θα καταγράφουν τις δικαιωτικέ και δικαστικέ αποφάσεις και θα περιλαμβάνουν τα μέτρα προστασίας υπέρ κάποια αδύναμου ατόμου, καθώς επίσης και ε, κάποια ε, εντολή αδυναμία. pour des raisons de confidentialité, de respect de la vie privée, de la sécurité juridique και θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται όσον αφορά την ασφάλεια δικαίου σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν ε, κατάλληλα μέτρα. Εάν υπάρχει κάποια επιβάρυνση, κυρίως για τη μεταφορά ενός ατόμου από τη μία χώρα στην άλλη, θα πρέπει να προβλέψουμε κάποιους μηχανισμούς ε, συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών των ε, ε, χωρών που άπτονται τη απόφαση και θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να κάνουν οι αρχές αυτές. Στόχος θα πρέπει να είναι η προστασία των συμφερόντων του αδύναμου ατόμου. Ολοκληρώνοντας, επιθυμώ η Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάστηκε 17 χρόνια να λύσει τα θέματα κληρονομικότητας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην χρειαστεί τόσο χρόνο για να ρυθμίσει τα θέματα των ευάλωτων ατόμων και ε, θα ήθελα επιτέλους να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό το ζήτημα χωρίς να υπάρχουν πολιτικές επιρροές ή οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, προσοχή σας. Λαμπρά, πιστεύω ότι θα εισακουστεί η ευχή σας. Ποιος θέλει το λόγο παρακαλώ, Τερέζα. Ευχαριστώ. Είμαι βέβαιη ότι όταν θα συζητήσουμε στην Επιτροπή τα ευάλωτα άτομα, είτε πρόκειται για παιδιά είτε για ενήλικες, ε, δυστυχώς ε, ακολουθούμε πολύ συχνά μια τακτική μικροκομματική. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε μια έκθεση, ε, οι συστάσεις της οποίας ε, αφορούν πράγματα γύρω από τα οποία υπάρχει ήδη εθνική νομοθεσία, η οποία είναι και πολύ ανομοιογενής και γνωρίζουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη πυκλομορφία νόμων σε εθνικό επίπεδο, αλλά το ζήτημα αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιληθεί ε, αν επιχειρήσουμε δηλαδή να τροποποιήσουμε ορισμένους από αυτούς τους εθνικούς νόμους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κάποιες συστάσεις που πιστεύω ότι αξίζει να υποστηριχθούν. Για παράδειγμα, ένα ε, θέμα που πρέπει πράγματι να τύχει της υποστήριξής μας ε, είναι ε, να παροτρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη-μέλη να ακυρώσουν τη σύμβαση της ε, Χάγης. Νομίζω ότι μπορούμε να ε, διευκολύνουμε την πρόσβαση στην, σε πληροφορίες και την προστασία των ευάλωτων ατόμων που χρειάζονται τις πληροφορίες. Και νομίζω ότι ε, υπάρχουν επίση τρόποι για τη βελτίωση της ε, συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της προστασίας των ευάλωτων ατόμων. Νομίζω ότι το πιο κρίσιμο σημείο σε αυτή την έκθεση θα είναι το πόσο ε, βαθιά μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς ταυτόχρονα να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη να τροποποιήσουν τη δική τους νομοθεσία για την προστασία των ευάλωτων ατόμων, κυρίως διότι πολύ συχνά η εθνική νομοθεσία βασίζεται και σε οικονομικούς, κοινωνικούς ε, παράγοντες και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του κάθε λαού και του κάθε πολιτισμού. Ε, εδώ ε, και, και, και μιλώ για την ε, δυνατότητα διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων από τα ευάλωτα άτομα αλλά και τη σχέση τους με, τα, με τους συγγενείς τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χάουταλα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Περζόν για το γεγονός ότι προσδιορίσε τόσες πολλές ε, κοινωνικές ομάδες που πράγματι ε, είναι ευάλωτες κατά τη μετακίνησή του από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσω και με αυτά που είπε η κυρία Κομοντίνη γιατί πράγματι αντιμετωπίζουμε, ε, υπάρχει μια τεράστια επικλομορφία ε, στις εθνικές νομοθεσίες και ε, προφανώς υπάρχει και αντίθεση από το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Το ερώτημά μου προς την Ζωή Μπερζερών είναι, λοιπόν, έχεις εντοπίσει ποια σημεία θα είναι τα πιο δύσκολα, θα είναι εκείνα γύρω από τα οποία θα ασκηθεί η μεγαλύτερη αντίσταση και, τα, και ποια θα είναι εκείνα τα οποία θα είναι πιο εύκολα ε, γιατί μόλις που κάνουμε τα πρώτα βήματα ως προς την κατανόηση του ε, συνολικού αυτού θέματος, ίσως θα έπρεπε να ακολουθήσουμε ε, μια πιο βαθμιαία προσέγγιση και να ακολουθήσουμε το παράδειγμα από άλλους τομείς πολιτικής, όπου ναι μεν όπως και εδώ υπήρχε ανάγκη αλλά όχι βούληση από τα κράτη-μέλη. Οπότε πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιες θα είναι συγκεκριμένα οι συστάσεις που θα κάνουμε εμείς. Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα με τις περισσότερες προτάσεις σας. Και εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να μιλούμε για τα θέματα αυτά σχετα με τη, την πολιτική μας ιδεολογία. Τους ε, τελευταίους μήνες στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, συζητάμε για πράγματα που υπάρχουν αλλά που δεν έχουν διαθετηθεί νομικά. Πιστεύω ότι και για αυτό το θέμα θα πρέπει να θεσπίσουμε κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, κυρίως ό,τι αφορά του ορισμού που καλό θα είναι να είναι κοινή. Γιατί το γεγονό ότι δεν υπάρχει κοινό ορισμό για τη συνήθη διαμονή, για τη δικαιοπρακτική ικανότητα αυτών των ατόμων. Ακριβώ επειδή υπάρχουν διαφορέ, έχουμε διαφορέ και στην εφαρμογή των προνομίων ή των διαφόρων ε, διατάξεων που ισχύουν για τα άτομα αυτά, που όμω μετακινούνται από μία χώρα σε άλλη. Και ακριβώ λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα θα πρέπει να ορίσουμε με κοινό τρόπο κάποια θέματα. Επίση για την εντολή μελλοντική προστασία, τα μέτρα προστασία. Ώστε από τη στιγμή που συμφωνούμε ότι υπάρχει μια κατάσταση θα πρέπει να τη ρυθμίσουμε και νομοθετικά. Ο μόνο μου προβληματισμός και η μόνη μου ανησυχία είναι να μην υποβάλουμε μια πρόταση εναρμόνισης που θα χρησιμοποιηθεί από τα κράτη-μέλη ως πρόσχημα για να αποφύγουν την εφαρμογή της ε, Σύμβασης της Χάγης. Θα πρέπει να δείξουμε στα κράτη-μέλη ότι μέσω της ε, πρότασής μας δίνουμε μια ευκαιρία σε αυτά για να ξεκινήσουν την εναρμόνιση σε ό,τι αφορά την ε, αντιμετώπιση των ευάλωτων ατόμων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφύγουν την κύρωση της Σύμβασης της Χάγης. Θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς εδώ. Ευχαριστώ κύριο Στουτιογόν. Ευχαριστώ. Καταρχήν, ω και ηγετής των Πρασίνων για το θέμα αυτό, θα ήθελα να υπενθυμίσω και πάλι στην κυρία Μπερζερόν ότι τη στηρίζουμε ανεπιφύλακτα στις προτάσεις της. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το ότι είναι πολιτικό αυτό το θέμα. Αλλά είναι πολιτικό με την πιο ευγενή έννοια του όρου. Θέλουμε να δώσουμε καρδιά στην Ευρώπη. Και για, να καταφέρει, αν καταφέρει η Ευρώπη να ε, εναρμονίσει οι εθνικές νομοθεσίες για τις τράπεζες, ε, για τις πολυεθνικές, αλλά δεν βρίσκει το θάρρος να ε, προκρίνει νομοθετικές ρυθμίσεις για να προστατεύσει ευάλωτα άτομα, ε, πώς δεν είναι πολιτικό αυτό το θέμα, αλλά με την πιο καλή έννοια, με την πιο ευγένεια. έννοια. Θα πρέπει επιτέλους ο άνθρωπος ε, να ε, υπερισχύσει της οικονομίας, ακόμη και των εθνικών διατάξεων. Ξέρω ότι δεν συμμεριζόμαστε όλη αυτή την άποψη, δεν πειράζει, και εγώ νομικός είμαι και πιστεύω ότι όταν η Ευρώπη προσπαθεί να προστατεύσει ε, τους αναξιοπαθείς, διαδραματίζει πραγματικά το ρόλο της. Δεν έχουμε φτάσει βέβαια ακόμη σε αυτό το στάδιο Ούτε κι εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμελήσουμε τη σύμβαση της Χάγης. Άλλωστε δεν είναι αυτή η πρόθεση ούτε της εισηγήτριας. Και θα πρέπει να, το αποφύγουμε, να αποφύγουμε οποιαδήποτε σχετική παρερμηνία. Πάντως οι πράσινοι στηρίζουν αμέριστα και με πυγμή την πρόταση της κυρίας Λεμπερζερό. Ευχαριστώ κύριο Σλιπρετό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα εγώ να σπείρω ζυζάνια ή να δημιουργήσω έρηδα, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει συνένεση, αλλά δεν είμαι τόσο ενθουσιώδης όσο εσείς για το θέμα αυτό. Σίγουρα το θέμα των ευάλωτων ενηλίκων είναι ένα σημαντικό θέμα που έχει και μέλλον, γιατί όντως το baby boom μετατρέπεται σε γέρο boom ε, και όλο πιο ευάλωτους ε, ηλικιωμένους έχουμε μεταξύ άλλων ευαλώτων. Και μάλιστα η Γαλλία πρόσφατα έκρινε νομοσχέδιο για την εντολή μελλοντική προστασίας. Καλό είναι το αποτέλεσμα γιατί έτσι μπορούν άνθρωποι που φοβούνται ότι θα γίνουν κάποια στιγμή ευάλωτοι, παρόλο που δεν είναι ακόμη ευάλωτοι, να βάλουν τα μέτρα τους για να οργανώσουν τη ζωή τους ώστε να μην ε, τους πιάσει απροετοίμαστη αυτή η κατάσταση να μην πιάσει στο συγγνώμη αυτή η κατάσταση. Πάντω, καλά ξεκινάει. Καλό είναι το σημείο αφετηρία τη κυρία Λεμπρετών, αλλά δεν καταλήγει σωστά. Γιατί ε, πολύ σωστά θα είναι τα κράτη-μέλη να κυρώσουν τη σύμβαση τη Χάγη που υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν να θαρρύνουμε τα κράτη-μέλη που έχουν ε, καθυστερήσει να την κυρώσουν. Βέβαια δεν περιορίζεται σε αυτό η συγγήτρια. Πάει ακόμη πιο μακριά και προτείνει έναν ευρωπαϊκό κανονισμό για το θέμα. Εκείνο που έχω πρόβλημα, καταρχήν και νομικό, γιατί υπάρχει ζήτημα επικουρικότητας εδώ και η αρχή της επικουρικότητας ε, δεν είναι εκεί για να τη βαραβιάζουμε, θα πρέπει που και που να τη σεβόμαστε και όλα. Επίσης υπάρχει και ένα ιονή φιλοσοφικό πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό το θέμα οφείλει να παραμένει στις εθνικές αρμοδιότητες. Βέβαια, επειδή υπάρχει και ένας διασυνοριακός χαρακτήρας, γιατί αυτοί οι ευάλωτοι ενήλικες μετακινούνται και όλα, θα πρέπει να επιλύσω αυτό το διασυνοριακό ζήτημα με μια ελαστική συνεργασία και όχι με ένα νομικά δεσμευτικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Φαίνεται ότι δεν ε, ε, διδαχθήκαμε ακόμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τα παθήματα του Brexit. Δεν είναι... Ε, δεν έγινε το Brexit επειδή ο Βρετανός Πάπας ήταν υπέρ της περισσότερης ολοκλήρωσης, αλλά ήθελα λιγότερη ολοκλήρωση. Και εμείς αντί να διδαχθούμε από το πάθημά μας, φαίνεται ότι οθούμε προς μεγαλύτερη ολοκλήρωση. Πραγματικά, αν δεν αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα, θα την πατήσουμε. Πάντως, εγώ σας προειδοποίησα. Πριν ξαναδώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν έχει κάποιες παρατηρήσεις. Ναι. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για την πλήρη έκθεσή και να υπενθυμίσει ότι το θέμα της προστασίας των ευάλωτων ε, ενηλίκων ε, το παρακολουθεί πολύ στενά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον από το 2008 όταν κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γαλλία κύρωσε την Σύμβαση της Χάγης για την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέτρεψε όλα τα κράτη-μέλη να την κυρώσουν αντιστοίχως. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία σε κάποιες από τις συστάσεις της έκθεσης και πιο συγκεκριμένα την σύσταση παριθμών 6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ήδη στα πλαίσια του Οικονομικού Προγράμματος Αστικής Δικαιοσύνης έχει συγχρηματοδοτήσει αρκετά ε, προγράμματα για την ε, ενημέρωση για την νομοθεσία όσον αφορά τους ευάλωτους ενήλικες, όπως για παράδειγμα το Συμβούλιο Συμβολογράφων ε, ε, της ε, Ευρώπης χρηματοδοτήθηκε η ιστοσελίδα τους. Υπάρχει μια ιστοσελίδα για τους ευάλωτους ενήλικες για θέματα μέτρων προστασίας για τους ευάλωτους αυτούς ενήλικες σε 22 ευρωπαϊκές χώρες. Και η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά. Όσον αφορά τη σύσταση υπαριθμών 7, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι η, Ευρωπαϊκή, η Επιτροπή Γιούρι είναι συνεχώς ενήμερη για τι δραστηριότητε που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Συμβουλίου προκειμένου να γίνεται ο απολαγισμός της κατάστασης για την κύρωση της ε, Σύμβασης της Χάγης του 2000 από τα κράτη-μέλη. Και το αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης ήταν ότι δεν υπήρχε ακόμα επαρκής εμπειρία προκειμένου να εκπονηθεί έκθεση επί του θέματος, διότι μόνο 7 κράτη-μέλη είχαν κυρώσει μέχρι σήμερα την σύμβαση και ακόμα και αυτά ε, ακόμα δεν έχουν ε, και τόση μεγάλη εμπειρία για την εφαρμογή της. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ενημερώσω και την Επιτροπή για το αποτέλεσμα της τελευταίας ε, διαβούλευσης ε, με τα κράτη-μέλη που είναι πάρα πολύ πρόσφατη διότι έγινε το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2016. Τα καλά νέα λοιπόν είναι ότι η Πορτογαλία, η Λετωνία και η Ιρλανδία ε, σκοπεύουν να κυρώσουν ε, εντός του έτους ε, τη σύμβαση, εντός του 2017. Η Σλοβακία ξεκινάει την προετοιμασία για την εσωτερική διαδικασία υπογραφής και κύρωσης της σύμβασης. Το Βέλγιο σκοπεύει να υπογράψει τη σύμβαση και θα ξεκινήσει τη διαδικασία κύρωσης μόλις έχει υπογραφεί η σύμβαση. Στην Ιταλία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την κύρωση της σύμβασης ε, είναι σε διαδικασία εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή στο Κοινοβούλιο. Και η ίδια κατάσταση ισχύει και στην Ελλάδα. Στη Σουηδία η έκθεση ε, του ερευνητή που διορίστηκε από την κυβέρνηση για να εξετάσει το θέμα της κύρωσης της ε, σύμβασης υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2015 και πρότεινε την κύρωση της ε, σύμβασης στην κυβέρνηση και η έκθεση και τα σχόλια από τις αρμόδιους φορείς τώρα εξετάζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Σουηδία. Αρκετά κράτη-μέλη ακόμα μελετούν τη σύμβαση ή ολοκληρώνουν την σε εσωτερικέ μεταρρυθμίσεις στην νομοθεσία τους όσον αφορά τους ευάλωτους ενήλικες. Η Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο για την Αγγλία και την Ουαλία, η Πολωνία, το Λουξεμβούργο, η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Δανία. Έχουμε ελάχιστες αρνητικές απαντήσεις. Η Κροατία και οι κάτω ε, έχουν δηλώσει ρητός ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να κυρώσουν τη σύμβαση λόγω του ε, μεγάλου δημοσιονομικού κόστους της εφαρμογής ε, της σύμβασης και η Ισπανία είπε ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για κύρωση. Δεν έχουμε ακόμα απαντήσεις από την Ουγγαρία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία, αλλά ε, τους έχουμε ήδη υποθυμίσει ότι πρέπει να μας στείλουν απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο ε, το συντομότερο δυνατόν. Η άποψη λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ε, σιγά σιγά αλλά σταθερά βελτιώνεται η κατάσταση και τα κράτη-μέλη όλο ένα και περισσότερο συνειδητοποιούν τη σημασία του ζητήματος. Το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει τη, στη σύσταση υπαριθμών οκτών αλλά λόγω της πρόσφατης αξιολόγησης που μόλις σας περιέγραψα, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η κύρωση της Σύμβασης της Χάγης. Στα πλαίσια της καλύτερης νομοθεσίας, που είναι μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επανάληψη του παρόντος νομοθετικού πλαισίου σίγουρα δεν αποτελεί μία από τις επιθυμητές μας επιλογές. Να επισημάνω επίσης ότι η μετάφραση της επεξηγηματικής έκθεσης προς την ε, ε, σύμβαση ε, σε όλες τις επίσημες γλώσσες που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα μέτρο για να προτρέψει τα κράτη-μέλη να την κυρώσουν, θα είναι έτοιμη τον Ιανουάριο. Ε, υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις γιατί επικαιροποιήθηκε το αρχικό κείμενο ε, του επεξηγηματικού κειμένου και γίνεται αναθεώρηση αντιστοίχω και των μεταφράσεων. Ε, επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει προετοιμασία για μια κοινή διάσκεψη με τη διάσκεψη της Χάγης κατά πάσα πιθανότητα του χρόνου στις αρχές του επομένου έτους ε, για το θέμα των ευάλωτων ενηλίκων και ε, πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη διάσκεψη θα αποτελέσει και μια ευκαιρία να ε, γίνει ανταλλαγή πρακτικών εμπειριών και έτσι να διευκολύνουμε και την κύρωση της σύμβασης. Βεβαίως θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε την Επιτροπή για την επόμενη διαδικασία κύρωσης το 2017. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχεις το λόγο για να ολοκληρώσουμε. Να ολοκληρώσουμε. Μα διαρωτώ με αν πραγματικά ακούσατε αυτά που είπα, Ζήλ και κύριε Κομοντίνη. Εγώ είπα ότι, ότι είναι ουσιαστικά αδύνατο να εναρμονίσουμε τις εθνικές νομοθεσίες. Και το μόνο που ζητήσαμε είναι η αναγνώριση της κατάστασης του ευάλωτου ατόμου και να μην υπάρχει ε, ανάγκη να ξαναγίνει αναγνώριση σε άλλο κράτος. Να μην χρειάζεται εκτελεστήριο τίτλος σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της κατάστασης της ε, ευπάθειας αυτής. Και ε, έχουμε διασυνοριακό χαρακτήρα. Ένα γαλλικό γάμο δεν αναγνωρίζεται στη Ρουμανία. Θέλουμε η κατάσταση ενό ατόμου να αναγνωρίζεται σε άλλο κράτο. Απλώ. Δεν ζήτησε να εφαρμοστεί ευρωπαϊκό δίκαιο ενιαίο σε όλα τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Παρά είμαστε σε πρώιμη φάση ανάπτυξη μα στην Ευρώπη για κάτι τέτοιο. Κάποια μέρα ίσω φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά δεδομένων των αντιστάσεων σε αυτή την πολύ μετριοπαθή ε, πρόταση που κάνω, βλέπω ότι ε, σίγουρα εμεί θα πεθάνουμε πριν φτάσουμε σε ένα θέμα αναγνώριση ε, ενό ευρωπαϊκού συστήματο δαιμονία για τέτοια θέματα. Ε, και σίγουρα είναι σωστή η ενθάρρυνση των χωρών μελών για την κύρωση, αλλά δεν είναι αποτελεσματικό το μέτρο. Το 2000 ε, υπεγράφει αυτή η συμφωνία. Έχουν περάσει 16 χρόνια και δεν έχουν κυρώσει οι χώρες ακόμη την σύμβαση αυτή. Πόσο να περιμένουμε, άλλα 20-30 χρόνια ε, θα πεθάνω. Δεν θα προλάβω να δω κάτι τέτοιο. Ε, γιατί αν πρέπει να περιμένουμε άλλα τόσα χρόνια, άλλα 30 χρόνια, καλά. Θα δούμε. Ελπίζω να είμαστε ακόμη εν ζωή όταν θα κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη αυτή η σύμβαση. Αν δεν κάνω λάθος, εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη. Διάφορα μόνο έχουν μείνει. Υπάρχει κάποιο σημείο για τα διάφορα? Όχι, οπότε... Επόμενες συνεδρίασεις... Να, έχασα το χαρτί. 24 Ιανουαρίου η συντακτική συνεδρίαση που θα κρατήσει μία ώρα και 30 και 31 Ιανουαρίου τακτική συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο.